να την πάρουν για παράδειγμα πολλοί από του συναδέλφου τη για την συμπεριφορά του εδώ στο σώμα. Ευχαριστώ. Ωραία. Τελειώνουμε τώρα τη συζήτηση για το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει την Τετάρτη το μεσημέρι. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη έκθεση, έκθεση της κυρίας Βένσον πλαίσιο πολιτικής της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Θα δώσω καταρχάς το λόγο στην κυρία Σβένσον ως εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους εισηγητές και το συναδέλφους στην Επιτροπή Ισότητας για την ε, δέσμευσή του όσον αφορά την καταπολέμηση βίας κατά των Ιρακών. ψηφοφορία, πριν από την ψηφοφορία της αύριο και τη συζήτηση, θα ήθελα να ξέρω πόσες γυναίκες αφορά αυτό. Πόσες γυναίκες δολοφονούνται, αλλά δεν θα το κάνω θα ήθελα να σας δώσω ορισμένες εικόνες από την βία αυτή για να τις έχετε κατά νου πριν από την ψηφοφορία ούτως ώστε κάθε βουλευτής να γνωρίζει ότι έχει τη δυνατότητα καταπολέμησης της βίας αυτής εάν υπερψηφίσει την έκθεση αύριο. Φανταστείτε, μια γυναίκα, μια μητέρα που διαβάζει μια ιστορία το βράδυ στα παιδιά της που έχουν μπει στο κρεβάτι Μπαίνει ο άντρα στο δωμάτιο και καταλαβαίνουν όλοι τι πρόκειται να γίνει. Τα παιδιά κρύβονται κάτω από την κουβέρτα, προσπαθούν να μην ακούσουν και να μην δουν τι γίνεται. Ακούν τον πατέρα να ουρλιάζει, ακούνε τον ξυλοδαρμό και ακούνε τη μητέρα να κλαίει και να αναστενάζει μία εικόνα αυτή, μια άλλη εικόνα. Μία γυναίκα η οποία πολλά χρόνια ζούσε θύμα βίας και αποφασίζει να φύγει από αυτή τη σχέση και να δημιουργήσει μια νέα σχέση, μια νέα ζωή με τα παιδιά της. Φεύγει. Έχει την τύχη να βρει μια θέση σε ένα οίκο προστασίας γυναικών και ο άντρα, όταν μετά από μέρες πάει τα παιδιά της στο νηπιογωγείο περιμένει ο πατέρας αυτός πριν έξω από το νηπιογωγείο ε, νηπιαγωγείο και την δολοφονεί, τη μαχαιρώνει. Και πεθαίνει γιατί είναι γυναίκα, για κανένα άλλο λόγο. Αυτή η θανατηφόρα βία κατά των γυναικών που μπορείτε να φανταστείτε γίνεται ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία η γυναίκα αυτή αποφασίζει να βγει από την ελόγω σχέση. Μια γυναίκα δεν μπορεί να πάρει διαζύγιο από έναν άντρα ο οποίος την θεωρεί ιδιοκτησία του και βρίσκεται σε μια κατάσταση τεραστίου κινδύνου γιατί ο άντρας καταλαβαίνει ότι χάνει την, ε, τον έλεγχο της γυναίκας αυτής. Μια άλλη εικόνα ένα κορίτσι ε, είναι στο σινεμά με κάποιο φίλο, φεύγει, λέει εντάξει τα λέμε αύριο, ακούει κάποιον να έρχεται από πίσω της, ο οποίος της επιτίθεται, τη βιάζει, επειδή μένει η κοπέλα, αλλά πρέπει όλη της τη ζωή να την περάσει με αυτό το τραύμα η Κομισιόν στο πρόγραμμά της, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, επιβεβαιώσει ότι το 2011-2012 θα ετοιμάσει μία ανακοίνωση για τις πράξεις αυτές βίας και θα πρέπει να υπάρχει και ένα πρόγραμμα δράσης σε κοινοτικό επίπεδο και χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα δράσης εφόσον οι γυναίκες υπόκεινται σε βία επειδή είναι γυναίκες δεν θα μπορεί κανένας να πει ότι ζούμε σε δημοκρατική κοινωνία, σε ισότιμη κοινωνία. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητες ε, ε, ζωής των γυναικών αυτών και πρέπει να μην ξεχνάμε πόσο διευρυμένη είναι η βία αυτή στην κοινωνία. Οι γυναίκες είναι θύματα αυτής της βίας που πλήττει το συγκεκριμένο φύλλο. Καμιά φορά πρέπει να ξεχνάμε να βλέπουμε τις γυναίκες μόνο σαν θύματα. Υπάρχουν και ισχυρές γυναίκε, οι οποίε με την υποστήριξη κοινωνία πετυχαίνουν να δημιουργήσουν μια καλή ζωή για τι ίδιες και τα παιδιά του. Και είναι έργο μα στο Κοινοβούλιο να δείξουμε ότι στηρίζουμε αυτέ τι γυναίκε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόκειται λοιπόν για την αντιμετώπιση των γυναικών που έχουμε. Η Επίτροπο, η κυρία Μάρστον, έχει το λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ κυρία Σβένσον για την πολύ συγκινητική εισαγωγή σας για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Η καταπολέμηση τη βίας κατά των γυναικών είναι υψηλή προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω δείχνει και η στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Όπως ε, είπατε κι εσείς, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα ε, βίας κατά των γυναικών στην Ευρώπη. Και για αυτό το λόγο ε, δουλεύουμε σε εστιασμένε δράσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Θα αναπτύξουμε μια σαφή πολιτική για να αντιμετωπίσουμε ακριβώ αυτό το πρόβλημα στην Ευρώπη. Καλωτοσορίζω την έκθεσή σας κυρία Σβένσον και αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία που πήρατε δίνει την ευκαιρία να ανταλλάσσουμε απόψει, να δημιουργήσουμε συνέργειε μεταξύ αυτού που κάνει η Κομισιόν και αυτού που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προσδιορίσουμε μελλοντική δράση για αυτόν τον τομέα. Ένα-δύο σημεία που αναφέρατε στην έκθεση καλύπτονται από τα προγράμματα δράση τη Κομισιόν για την καταπολέμηση τη βία εναντίον των γυναικών. Για να ενισχύσουμε την επίδρασή μας, ε, εστιάζουμε συγκεκριμένε δράσει όπου υπάρχει συγκεκριμένη νομική βάση με βάση συνθήκη τη Λισαβόνα. Στο πακέτο για τα δικαιώματα των θυμάτων που θα ετοιμαστεί, θα αντιμετωπίσουμε ειδικά τα θύματα των ιδιαίτερα ευάλωτων ανθρώπων, όπως των γυναικών και των παιδιών. Το πακέτο αυτό θα παρουσιαστεί τον επόμενο μήνα. Κάθε εβδομάδα τα θύματα αυτά χρειαζόνται βοήθεια ε, μετά από την επίθεση που τους ε, έχει γίνει. Οι γυναίκες φυσικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτες εφόσον έχουν πληγεί από βία κατοίκων, βιασμό ή σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή βίας. Θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε με σεβασμό και με γνώση ε, κατά τις επαφές τους με τους ανθρώπους το σύστημα δικαιοσύνη. Θα πρέπει να τι υποστηρίζουμε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και στη δικαιοσύνη και σε αποζημίωση. Το νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπει ένα ελάχιστο επίπεδο αποζημίωση για τα θύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξάρτητα με τον τόπο που έπεσαν θύματα. Γι' αυτό η Κομισιόν θέλει να δράσει και να ενισχύσει τη θέση των θυμάτων στην Ευρώπη. Θα παρουσιάσει λοιπόν ω πρώτο βήμα ένα πακέτο ε, νομοθετικών μέτρων για τα δικαιώματα, την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων αδικημάτων και την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασία. Ε, συγκεκριμένη εστίαση θα δοθεί σε ευάλωτα θύματα όπως θύματα σεξουαλικής βίας και οικιακής βίας. Η Κομισιόν θα υποστηρίξει επίσης μέτρα προστασίας αμοιβαίας αναγνώρισης που θα ωφελήσουν κυρίως ε, θύματα που έχουν πέσει κατ' επανάληψη θύματα των συζύγων τους, μελών της οικογένειας κτλ. Με το πακέτο αυτό η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ότι στην Ευρώπη καμία γυναίκα που θα περνάει τα θύματα και δεν θα, υποφελεί, δεν θα ξεφεύγει από το μηχανισμό προστασίας ε, στα πλαίσια του ποινικού και αστικού ε, συστήματος. Το πακέτο αυτό θα συμπληρωθεί με άλλα μέσα που θα εστιάζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάποιων ειδών θυμάτων. Φερρυπίν, η Κομισιόν θέλει να αναλάβει ισχυρή δράση για να καταπολεμήσει ε, τον ακροτηρισμό των γυναικείων ε, σεξουαλικών οργάνων. Παράλληλα ε, με τις δράσεις μας στον ποινικό τομέα θα ενισχύσουμε τη θέση των γυναικών, θα υπάρξει αφύπνισή τους και θα αναλύσουμε τις στατιστικές για τη βία που υφίστανται. Η Κομισιόν θα βασιστεί στη δουλειά που, έκαναν, που έκανε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων θα, που συλλέγει και αναλύει τι στατιστικέ για το θέμα αυτό. Καταλήγοντα, θέλω να τονίσω ότι η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δίνει σημαντική οικονομική στήριξη για να προλάβει και να καταπολεμήσει τη βία μέσω του προγράμματο Δάφνη, Δάφνη δηλαδή 3, μέσω τη δουλειά που κάνει και τη συνεργασία με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει επίση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε, κυρία Επιτροπέ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο ή στους συναδέλφους από πλευράς των πολιτικών ομάδων. Και πρώτα πρώτα για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μπεσερίλ Τερίζο και Σχημένεθ Μπεθερίλ. Eh, η κυρία Χιμένεθ Μπεθερίλ, σας ευχαριστούμε. Τις περισσότερες φορές που έχω λάβει το λόγο εδώ στην Ολομέλεια το έκανα για να καταγγείλω τη βία κατά των γυναικών. Και εκ νέου είμαι εδώ για να καταβολήσω αυτό το φαινόμενο διότι θα πρέπει να σας πω ότι δεν με κουράζει να το κάνω αυτό συνέχεια, διότι θεωρώ ότι είναι απαραίτητο δημοσία να καταγγέλουμε αυτή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα υπέρ αυτής τη συμπεριφορά και νομίζω ότι αυτό που έχω στη διάθεσή μου είναι το βήμα αυτή τη ολομέλεια για τι γυναίκε εκείνε οι οποίε κάθε μέρα τις χειρίζονται και που χρειάζονται εμείς οι νομοθέτε, να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τι κυρώσει σε αυτού που του επιτίθενται διότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα αλλά επίση θα πρέπει να κάνουμε κάτι και για να πλαισιώσουμε τα ε, θύματα γιατί έχουμε όλε αυτέ τις, τις ε, τέταρτον περίπου των γυναικών που έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του αυτού του είδου τη βία ε, επίσης αυτό αφορά και ανήλικες. Όμως επομένως πρέπει όπως είπε και η Κομισιό να αναλάβουμε δράση, να δεσμευτούμε πέρα αυτής της πρωτοβουλίας και οπότε γι' αυτό και χρειάζεται ε, να, να επιμείνουμε σε αυτή την ερώτα και πάλι να προστατεύσουμε αυτά τα θύματα γιατί άλλωστε είχα κάνει και αυτή την εισήγηση και οπότε θα πρέπει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία επιψηφίσαμε να γίνουν πραγματικότητες γιατί θυμάμαι ότι είχε υπάρξει μεγάλη συνένεση για την πρότασή μου οπότε θα πρέπει να δούμε ότι για να καταπολύσουμε την υγειακή βία είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τους πάντες, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, γυναίκες και άντρες οπότε δεν θα πρέπει αυτό να είναι αντικείμενο μικροπολιτικής και οπορτουνισμού και επομένως θα πρέπει αυτού του είδους την κοινωνική πληγή να την καταπολεμήσουμε όχι στην ε, ένοχη σιωπή εδώ και ε, δεκαετίες μιλούμε για την ε, βία των γυναικών αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι για να μειωθούν τα θύματα. Επομένως κάτι πάει στραβά και ήρθε τώρα η ώρα να αφήσουμε στην άκρη τη δημαγωγία και να μπορέσουμε από τα λόγια προχωρήσουμε στις πράξεις και επομένως θα πρέπει να υπάρξει κάποια ουσιαστική βοήθεια, ουσιαστική εφαρμογή του δικαίου για να μπορέσουν με αξιοπρέπεια να ζήσουν οι γυναίκες και με ασφάλεια. Και όλα τα δήματα να ξέρουν ότι εγώ θα είμαι εδώ και θα υψώνω τη φωνή μου ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το, το, το, τέρας το, το οποίο κοστίζει τόσες αθώες ζωές. Φτάνει πια και ελπίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Και δεν θέλω να διακόψω, ε, αλλά θα πρέπει να σας παρακαλέσω για άλλη μια φορά να τηρείτε τα χρονικά ώρα. Έχετε 1,5 λεπτό για το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Η κυρία Τόμσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μία στις δέκα γυναίκες έχει υπάρξει θύμα αυτής της βίας. Άρα και πολλοί ανήλικοι έχουν υποστεί σωματική βία. Στην Ευρώπη γίνονται αυτά. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι δυνατόν να κλείνουμε τα μάτια σε αυτή την πραγματικότητα. Ούτε θέλω κανείς να μου ξαναπεί παραμύθια για το βιτριόλι και τα οξέα και όλα αυτά που, που τους πετάνε για να τις παραμορφώσουν οι σύζυγοί τους. Πρόκειται για ένα σκάνδαλο. Θα πρέπει σε Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να κάνει για να βάλει φρένο σε αυτή την βία. Οπότε θα πρέπει να λέμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια έκθεση πάρα πολύ ε, σημαντική. Είναι ένα μήνυμα προ τον έξω κόσμο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι η βία των γυναικών είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένω, θα πρέπει να λάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζεται μια οδηγία. Μια οδηγία ούτω ώστε να σταματήσει η βία. Και χρειαζόμαστε επομένω να συντονιστούμε όσον αφορά την προσέγγιση μα και να εξασφαλίσουμε ότι τα βήματα θα προστατεύονται όσο γίνεται περισσότερο και ότι δεν θα υπάρξει περισσότερο αυτή η βία. Πρόληψη, πρόληψη χρειάζεται. Γιατί δεν είναι η ιδιωτική υπόθεση αυτή. Δεν είναι τα κατοικοθά. Επομένω θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να σταματήσουμε. Σα παρακαλώ τώρα πάρα πολύ να λάβετε το λόγο για του ε, δημοκράτε, φιλελευθέρου. Η επόμενη συνάδελφο που είναι η κυρία Παρβανόβα και έχει το λόγο δια δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι θα πρέπει να συγχαρούμε την εισηγήτρια για το έργο το οποίο επετέλεσε και θα πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί κάτι για να σταματήσει η βία των γυναικών. Με αυτή την έκθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι άμεσα χρειάζεται να ληφθεί δράση για να καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απλώ αναγκαίο, είναι κατεπήγον. Θα πρέπει να συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα τα επιχειρήματα κατατείνουν στο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί παν μέτρων απαραίτητο, διότι γνωρίζουμε ότι ε, ε υπάρχει νομοθεσία στα κράτη-μέλη ε, αλλά χθες έγινε, ε, έγινε μια μελέτη βιωσιμότητας που λέει ότι οι υπηρεσίες πλαισίωσης, οι εμπειρογνώμονες, οι, οι δυνατότητες των, των κρατικών υπηρεσιών δεν επαρκούν γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει βία κάθε μορφής και χρειάζεται σε ενωσιακό επίπεδο ένα, ένα πλαίσιο και να μην ξεχνούμε αυτό το χάρτη ε, που παρουσιάζεται πέρσι σε συνέχεια του προγράμματος τη Στοκόλμης Όμω παρόλα αυτά τα κράτη-μέλη δεν τα κατάφεραν όλη τη σχετική νομοθεσία να την ε, υλοποιήσουν για να προστατεύσουν την ε, γυναίκα για δυσμενεί διακρίσεις αλλά και βία. Διαπιστώνουμε επομένω τώρα ότι αδυνατεί να προστατεύσει του μισού πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, θα πρέπει η Κομισιόν τώρα να κάνει μια ad hoc νομοθετική πρόταση, να βάλει κάποιο ελάχιστα προαπαιτούμενα και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν νόμος και έτσι να έχουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική και να καλύψουμε πάσα μορφή βία και των γυναικών. Επομένω, χρειάζεται ε, πρωτοβουλία, χρειάζεται στρατηγική. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμο τι γίνεται με διάφορε δραστηριότητε και ίσω θα πρέπει να υπάρχει και μια χρονιά καταπολέμηση τη βία και των γυναικών στην Ευρώπη. Ε, γι' αυτό μαζεύουμε υπογραφέ των ε, πολιτών. Ε, άλλωστε πρόκειται και για θεμελιώδεις αρχές που ενσωματώνονται στην συνθήκη. Άρα θα πρέπει ξεκάθαρη απάντηση να, να δώσετε σήμερα πώς και πότε θα προτείνετε αποτελεσματικά μέτρα. Ευχαριστώ. Κυρία Παρβάνοβα, τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Κορνελίσεν από τους Πράσινους. Έχετε 1,5 λεπτό. Ε, I am happy that... Χαίρομαι που η καταπολέμηση τη βία βάσει του φύλου λόγω του φύλου είναι προτεραιότητα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κοινό ο στόχο αυτό, λοιπόν, για να υπάρξει πραγματική πρόοδο τα επόμενα χρόνια. Ελπίζω η έκθεση αυτή θα θεωρηθεί μια σημαντική συνεισφορά για το πακέτο των θυμάτων που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα υποσχέθηκε. Και το πακέτο αυτό για τα θύματα, με τη σειρά του, θα είναι μία από τι πτυχέ μια πανευρωπαϊκής στρατηγικής που θα συμπεριλαμβάνει υποστήριξη προ τα θύματα αλλά και άλλα ζητήματα ε, σε αυτόν τον αγώνα κατά πολέμηση του φαινομένου. Χρειαζόμαστε, Φερρυπίν, ένα ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών προστασία. Κάθε γυναίκα θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε καταφύγια, σε δωρεάν νομική βοήθεια και σε ψυχολογική βοήθεια. Φερρυπίν, χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε και τι μετανάστριε, οι οποίε δεν έχουν ε, μια ανεξάρτητη ε, άδεια κατοικία και είναι ιδιαίτερα ευπαθή. Αυτή η έκθεση έχει πολλά σημαντικά στοιχεία και ως πράσινοι ελπίζουμε ότι θα υπερψηφιστεί αυτή η έκθεση και θα την υπερψηφίσουμε και εμείς. Αν η παράγραφος 19 και το εκτιμώντα J παραμείνει που θεωρεί ότι η πορδία είναι παραβίαση των ε, θεμελιωτών δικαιωμάτων χωρίς να κάνει διάγραση ανάμεσα στην ε, εθελοντική και τη μη εθελοντική πορνεία, εμείς θα απόσχουμε. Ελπίζω να μην φτάσουμε εκεί και ελπίζω να υπάρξει μια ευρεία συνένεση υπέρ της έκθεσης ε, που θα την απευθύνουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς τα κράτη-μέλη και θα είναι η δική μας ξεχωριστή συνεισφορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Τσέσκοβα έχει το λόγο δύο-δύο λεπτά εκ μέρου των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαιρετίζω αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν νομοθετικά μέτρα για να υπάρξει ανάσχεση αυτού του φαινομένου της βίας εναντίον των γυναικών. Μία ε, σημαντική μορφή βίας είναι η βία στο σπίτι. Η βία αυτή στο σπίτι δεν είναι ιδιωτική υπόθεση της οικογένειας. Η ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών δεσμεύεται να υποστηρίξει τις οικογένειες και κυρίως τα παιδιά. Αυτό συνδέεται, αυτό το φαινόμενο είναι η βία στο σπίτι, η οικιακή βία και έχει καταστροφικές συνέπειες για όλα τα μέλη της οικογένειας, ιδίως για τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία γίνονται μάρτυρες αυτής της βίας στο σπίτι τους με τρόπο επαναληπτικό και θεωρούν τη βία ως ε, κάτι το συνηθισμένο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν στο μέλλον και τα ίδια τα παιδιά αυτά ως ενήλικες θα γίνουν βίαιοι άνθρωποι. Η βία εναντίον των γυναικών ενισχύει κατά την γνώμη μου την ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και επηρεάζει τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Οι γυναίκες οι οποίες υφίστανται οικιακή βία συχνά είναι και οικονομικά εξαρτημένες από το δράστη, από τον ένοχο αυτής της βίας. Θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες για να αποκαλύψουμε αυτά τα περιστατικά βίας και θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στις κοινωνίες μας για το φαινόμενο αυτό. Θα πρέπει να υπάρξουν ε, επίσης ενημερωτικές εκστρατείες για το φαινόμενο αυτό, γιατί συχνά οι γυναίκες διστάζουν να μιλήσουν δημόσια για τις εμπειρίες τους. Τα νομοθετικά μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο Παραδείγματο χάρη, ε, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη για τα θύματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν πολύ. Η κυρία Φιγκερέιδο τώρα. Από την ε, αριστερά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μια πολύ σημαντική έκθεση που μας προτείνει να αντιμετωπίσουμε σφαιρικά, ε, με πολιτικό τρόπο, αυτό το φαινόμενο της βίας λόγω Μιλάμε για συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν ε, έως και τις ε, ποινικέ διαδικασίες, αλλά και προληπτικά μέτρα και μέτρα προστασίας. Μας τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε συγκεκριμένες ε, προϋποθέσεις για τη χειραφέτηση των γυναικών. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την ενέργεια την τη δουλειά η οποία δεν είναι σίγουρη, τη φτώχεια, ούτως ώστε οι γυναίκες να επιλέγουν ελεύθερες με ποιο τρόπο θέλουν να ζήσουν. Δυστυχώς αυτό σήμερα δεν συμβαίνει. Και πολύ συχνά οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να ζήσουν ε, μέσα σε συνθήκες εξάρτησης ή θα πρέπει να ε, αναγκαστούν, εξαναγκάζονται σε πορνεία ή πέφτουν θύματα οικιακής βίας κτλ. Μιλάμε για καταστάσεις ε, που δεν επέλεξαν σίγουρα αυτές οι γυναίκες. Είναι η στιγμή να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις και να θέσουμε τέρμα σε αυτή τη βία, που είναι μία από τις πιο σοβαρές μορφές παραβίασης των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δεχόμαστε αυτή την συγκεκριμένη βία που βασίζεται στο φύλλο, που έχει τρομακτική επίπτωση και στα παιδιά και που επιδεινώνεται σε μια στιγμή κοινωνική και οικονομική κρίση. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να παρέμβει το συντομότερο δυνατόν, αλλά και τα κράτη-μέλη επίση θα πρέπει να κάνουν και αυτά ό,τι μπορούν με συγκεκριμένα μέτρα για να υπερασπιστούν τι γυναίκε. Πρόεδρο. Τώρα. Οι μεμονωμένοι ομιλητέ θα πάρουν το λόγο. Καταρχά η κυρία Ματέρα έχει δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η καταπολέμηση όλων των μορφών βίας ε, εναντίον των γυναικών είναι μία από τις προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητάω λοιπόν να υιοθετηθούν μέτρα μακροπρόθεσμα στον τομέα τον πολιτικό, τον κοινωνικό και τον ε, ε, δικαστικό, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτή τη βία λόγω φύλου και να φτάσουμε σε μια πραγματική ισότητα μεταξύ των φύλων. Εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθήσαμε ε, την ιδέα της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού έτους ε, για την καταπολέμηση αυτής της βίας με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Η αναγνώριση αυτού του σχεδίου δράση από, Ευρωπαϊκής Επιτρο... Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση αυτής της βίας 2010-2015 θα πρέπει να μεταφραστεί συγκεκριμένα μέτρα. Περιμένουμε ακόμα το στρατηγικό σχέδιο που μας εξαν... εξήγηλε η Επιτροπή για φέτος. Θα υπάρξουν δηλαδή, μας είπε, ε, νομοθετικά και πρακτικά μέτρα, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε στα θύματα την κατάλληλη προστασία ε, στα πλαίσια των εθνικών συστημάτων, ε, στα πλαίσια πιο συγκεκριμένα της ποινική δικαιοσύνης. Εκτιμούμε ότι μεταξύ του 20 έως από 20 με 25% των γυναικών στην Ευρώπη έπεσαν θύματα τουλάχιστον μία φορά της, ε, στη ζωή τους θύματα. Ε, και μισέ, μισό εκατομμύριο γυναίκες έπεσαν θύματα ακροτηριασμού των ε, οργάνων τους, των γεννητικών οργάνων τους. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικά φαινόμενα και θα πρέπει πάρα αυτά να παρέμβουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η βία κατά των γυναικών έχει τεράστια, τεράστιες και καταστρεπτικές συνέπειες στις γυναίκες. Οι μητέρες δεν μπορούν πια να εξασφαλίσουν την ασφάλεια στα παιδιά και τα παιδιά γίνονται έμεσα θύματα αυτής της βίας. Η βία εναντίον των γυναικών είναι ένα φαινόμενο πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε, γιατί πολύ συχνά οι ίδιες οι γυναίκες, στα θύματα, ντρέπονται και φοβούνται να καταγγείλουν στις αρχές την ε, βία που, που υφίστανται. Τώρα, καταλήγω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το έργο των θεσμικών οργάνων, αλλά είναι και απαραίτητο. Ε, και εγώ θέλω να πω Τέλος αυτή τη βία εναντίον των γυναικών, τέλος αυτή τη στιγμή, όχι αύριο. Εστρέλα και Και τώρα έχει το λόγο η κυρία Εστρέλα. Έχετε ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια και δεν μπορώ παρά να συγχαρώ την εισηγήτρια για το αξιόλογο αυτό έγγραφο το οποίο οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες θα επιψηφίσουν. Είπαν οι προλαλήσαντες και προλαλήσασες ότι η βία των γυναικών αποτελεί μια σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι γνωστό ότι τα θύματα της βίας αυτής υποχρεούνται να απεμπολίσουν πολλά τους δικαιώματα και επομένως έτσι είναι ευάλωτες σε μια εκ νέου άσκηση βίας. Έχω δουλέψει χρόνο την Πορτογαλία με γυναίκες τέτοιες που έχουν πέσει θύματα αυτού του φαινομένου και ε, μίλησαν για μια ζωή γεμάτη βάσανα. Και μόνο υπό την πίεση των παιδιών τους πήγαν και κατήγγυλαν αυτούς που τις χτύπησαν. Σε άλλη περίπτωση δεν είχαν το θάρρος να πάνε να κάνουν την καταγγελία, οπότε τα παιδιά πηγαίνουν και την έκαναν για αυτές. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει κάπως να βγουν αυτές οι γυναίκες, να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, να πάρουν τα παιδιά τους μαζί τους για να αφήσουν ε, αυτόν που τους επιτέθηκε στο σπίτι. Μόνο τους. Άρα θα πρέπει κάποιο, τρόπο να εξασφαλίσουμε το να έχουν αξιοπρέπεια οι γυναίκες, να σταματήσουν να είναι θύματα βίας. Να σταματήσει αυτό το φαινόμενο κατά το οποίο οι γυναίκες πέφτουν θύματα τέτοιων καταστάσεων που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από κανένα. Επομένως να λάβετε υπόψη ότι πρόκειται εδώ πέρα ουσιαστικά για υπονόμηση της δημοκρατίας. Γιατί οι γυναίκες που έχουν υποστεί τέτοιες ε, επιθέσεις δεν έχουν πια το δικαίωμα που έχουν όλοι οι πολίτες σε μια δημοκρατία. Άρα όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε να το σταματήσει το φαινόμενο. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και έχει τρώτο λόγο ο κύριος Κόφσκι. Να, να μιλήσει και ένας άντρας ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη εικόνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βία κατά των γυναικών, βία που ασκείται στο σπίτι. Φένσον. Θα πρέπει να ζαληθούν μέτρα σε νομικό επίπεδο. Άρα, συμφωνώ με την κυρία Σβένσον, όμως εγώ θα καταγγείλω και άλλη μία μορφή βίας. Η βία που υφίστανται οι γυναίκες από το κράτος, το κράτος που τους αρπάζει τα παιδιά τους. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Αυτή είναι η χειρότερη βία που μπορεί να υποστεί μια γυναίκα, το να της πάρουν το παιδί της. Αυτό γίνεται πολλές φορές με δικαστική απόφαση. Ένα δεκάχρονο πήραμε από το παιδί του πρόσφατα. Και είπαν ότι η γυναίκα του, η, η μάνα του παραπροσεύχεται. Και πολλές φορές αυτό το κάνουν για λόγους κακής οικονομική κατάστασης. Δεν να βοηθήσουν οικονομικά τους γονείς, παίρνουν το παιδί και το πάνε σε ορφανοτροφείο. Και τα παιδιά αυτά πολλέ φορέ, πάνε και τα παίρνουν επειδή υπάρχουν προστριβές και καβγάδες μέχρι των γονέων. Άρα θα πρέπει να αναλυφθεί δράση κατά αυτόν τον φαινομένων γιατί πώς η αστυνομία ή άλλου είδους δημόσιες αρχές προβαίνουν σε αυτή την πράξη. Έχουμε τάση αυτή να υποτιμούμε την οικογένεια και αν θεωρούμε ότι η κρατική παρέμβαση στο βωμό κάποιου νόμου τα δικαιολογεί όλα. Έτσι, στερείται η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν δικαιολογούνται αυτά. Με τίποτα. Οι φτωχοί θα πρέπει οικονομικά να στηρίζονται, αλλά δεν είναι δυνατόν οι οικογενειακοί δεσμοί να θράβονται έτσι βία. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κυρία Σκριδεύσκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια αυτής της Ολομέλειας το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μία έκθεση που μιλάει για το πολυσχηδές φαινόμενο του, του, της βίας κατά των γυναικών. Ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε την καταπολέμηση αυτού του αρνητικού φαινομένου. Φυσικά μόνο μια σφαιρική προσέγγιση σε πολλά επίπεδα, πολιτικό, κοινωνικό, νομικό, εκπαιδευτικό, μπορεί να δώσει οποιαδήποτε αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ότι μια πρόταση οδηγίας ε, που θα εστιάζει στην καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών που θα μας ετοιμάσει σύντομα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει. Έχω και άλλες παρατηρήσεις να κάνω. Αυτή η βία εναντίον των γυναικών θα πρέπει να θεωρείται όχι μόνο κάτι κακό για τις ε, γυναίκες ή για την ε, οικογένεια, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε το κόστος για όλη την κοινωνία αυτού του φαινομένου. Η συζήτηση τώρα για αυτό το θέμα δεν θα πρέπει να αφορά μόνο την καταπολέμηση της βίας αυτής καθεαυτής, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και κάποια ε, μοντέλα συμπεριφοράς η αποδοχή της βίας θα πρέπει να στιγματίζεται. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι επιπτώσεις έχει, πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε αυτά τα σπίτια, τι ποιότητα ζωής έχουν στην καθημερινότητά τους. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που παρουσίασε μια τόσο σημαντική έκθεση και πιστεύω ότι μετά τη σημερινή συζήτηση θα σταματήσουμε να μιλάμε μόνο για τη βία εναντίον των γυναικών, αλλά θα αρχίσουμε να ε, λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των γυναικών. Ευχαριστώ. Ο επόμενο ε, είναι η κυρία Μποσκούρτα. λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης, η Κομισιόν Μα είπε ποια είναι όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταπολεμήσουμε την δία εναντίον των γυναικών. Παρ' όλα αυτά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια στρατηγική σφαιρική. Ε, κάτι που το χρειαζόμαστε όμως, και είναι εκ των όνων Καλή ασφάλεια, Ιδίω για τους πιο ευπαθείς μεταξύ ημών. Για τόσε γυναίκες, α πούμε, οι οποίε είναι θύματα μέσα σε γάμου που δεν του διάλεξαν, γυναίκε που πέφτουν θύματα γιατί τους ακροτηριάζουν τα γενετικά τους όργανα. Ε, πάρα πολλές κοπέλες στην Ευρώπη πέφτουν θύματα αυτής της βίας. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά πρέπει να κάνουμε και έρευνε, να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή για τα θύματα αυτών των πρακτικών. Η Κομισιόν θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να μα παρουσιάσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε τη βία αυτή. Μια στρατηγική που θα καταπολεμάει και αυτές τις παραδοσιακές πρακτικές. Το 2011 είναι απαράδεκτο ε, να μην έχει τεθεί σε ε, να μην έχουν τεθεί σε ισχύ, ας πούμε, ε, συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των γυναικών. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Σιμάσκι δεν είναι μέσα στην αίθουσα από ό,τι βλέπω. Αν είναι όμως του δώσω το λόγο για δύο λεπτά. Σε σχέση με αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ε, και η κυρία Σβένσον, η συγγήτρια, θα ήθελα να σας πω ακόμα μια φορά ότι η βία ε, ε, κατά των γυναικών αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Μία από τις αιτίε είναι η χαμηλή θέση των γυναικών, οι οικονομικές διακριτικές διακρίσεις και χαμηλότερη πρόσβαση σε θέσεις απασχόληση, χαμηλότερο μισθός και χαμηλότερο κοινωνικό στάτου από τι γυναίκες. Κι όμως, οι γυναίκες φέρουν το βάρο της ανατροφή των παιδιών. Και πολλέ ευρωπαϊκές χώρες δεν τις προστατεύουν επαρκώς. Ε, έχουμε ασθενή κοινωνικά μέτρα. Ε, και με αυτόν τον τρόπο εξασθενούμε τι γυναίκε και τι καθιστούμε ε, εξαρτώμενα μέλη από του συζύγου του. Αυτή η κατάσταση δεν είναι σωστή και δεν πρέπει να συνεχιστεί. Θα πρέπει να τις ανταμείψουμε για το χρόνο που αφιερώνουν για τη μητρότητα και την άτροφη των παιδιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα. Τη στιγμή που η Ευρώπη έχει τέτοιες οικονομικές δυσκολίες λόγω της δημογραφικής της κατάστασης αν υπήρχαν επιδόματα θα βοηθούσαν τις γυναίκες και νομίζω ότι θα τις προστάτευαν και θα τις θωράκιζαν σε κάποιο βαθμό εναντίον της βίας. Η εξάρτηση οικονομική των γυναικών από τους συζύγους τους είναι μία από τις παθητικότητάς τους και μία από τις αιτίες που τις καθιστά ευάλωτες. Και γι' αυτό το λόγο ανέχονται αυτή τη θέση του θύματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να βελτιώσει την κατάστασή τους. Ιδίως ε, σε χώρες όπου η θέση των γυναικών είναι πολύ δύσκολη λόγω φτώχεια. Γι' αυτό ε, θέλω να περάσει αυτό το σημαντικό μήνυμα. Ε, είμαι ευγνώμων προς, τον, ε, προς την εισηγήτρια που σημείωσε αυτό το πρόβλημα και υπέδειξε και τη λύση. Ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Εντίτ Μπάουερ για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τόσο καλή αυτή τη έκθεση. Θεωρώ ότι πραγματικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό θέμα. Στην Ευρώπη έχουμε συνηθίσει πολλά να γίνονται. Όταν λέμε ότι κάποιο θέμα έχει οικονομική σημασία. Αυτή η έκθεση όμως καταδεικνύει ότι ε, δαπανούνται δισεκατομμύρια κάθε χρόνο ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτά τα θύματα, τις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Η βία αυτή είναι όλα τα επίπεδα. Αφορά και φτωχούς και ε, πλούσιους, μορφωμένους και αμόρφωτους. Εκατοντάδες γυναίκες κάθε χρόνο είναι θύματα της οικογενειακής βίας. Στην Ευρώπη έχουμε διαφορετικές μορφές της βίας αυτής κατά των γυναικών, εκτός των οποίων ορισμένες ήδη αναφέρθηκαν. Αναφέρθηκε επίσης ότι οι γυναίκες χάνουν την αυτοπεποίθησή τους αν είναι θύματα βίας, ότι δεν ελέγχουν πια την ίδια τους τη ζωή. Και ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πραγματικά μια νομική βάση αντίδρασης. Μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Ακόμα και αν δεν είναι αρρωσμένα τα διάφορα νομικά συστήματα στα κράτη-μέλη, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Έστω και μια ανταλλαγή απόψεων. Ήδη και αυτό βοηθά. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι υπάρχουν εγκλήματα ε, τα οποία σε ορισμένες χώρες όμως δεν καλύπτουν τη βία κατά των γυναικών. Εκεί πρέπει να δράσουμε, εκεί πρέπει να συνεργαστούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγία κατεπηγόντως. Ευχαριστώ και Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια την κυρία Σβένσον. Η βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση που μας την υποσχέθηκε ε, για μια στρατηγική καταπολέμησης ε, της βίας που θα είναι σφαιρική. Θα αφορά και την οικιακή βία και τον ακροτηριασμό των γυναικείων οργάνων αλλά και άλλες μορφές βίας. Μιλάω ε, για την παρενόχληση ας πούμε ε, των εργαζόμενων γυναικών ή παραδείγματο χάρη την παρενόχληση των εγγύων γυναικών στον χώρο εργασία που τις εξαναγκάζουν σε παρέτηση ή παραδείγματο χάρη ε, τη θέση και τον τρόπο που παρουσιάζονται οι γυναίκες στην τηλεόραση και στη διαφήμιση. Η Επίτροπος η κυρία Μάλστρομ μας εξήγηλε μέτρα υπεράσπισης των θυμάτων. Θα πρέπει να υπάρξει ε, μεγαλύτερη εναρμόνιση των κανόνων και αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών τη σημασία των αδικημάτων αυτών. Ε, και επίσης όταν τα θύματα είναι ανήλικες γυναίκες είναι ειδική κατηγορία. Θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη προστασία, προξενική προστασία, συνεργασία με μη κυβερνητικέ οργανώσει, συνεχείς ε, στατιστικέ συγκρίσιμε, ανάλυση επιπτώσεων για να δούμε ε, με ποιου τρόπου μπορούμε να προλάβουμε το φαινόμενο αυτό στα κράτη-μέλη και τι κάνουν τα κράτη-μέλη για να υπάρξει συγκεκριμένη μείωση του φαινομένου. Νομίζω ότι υπάρχει κοινή θέληση του Κοινοβουλίου και εγώ προσυπέκλεψα την ε, δήλωση αυτή για να προβλέψουμε ένα έτος όπου θα προβληματιστούμε για το φαινόμενο αυτό σε όλη την Ευρώπη. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο ε, η φωνή μας θα είναι πραγματικά ηχηρή και θα μας ακούσουν όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μπάστος για δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι, πρόκειται εδώ πέρα για κάποια πάρα πολύ σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και αυτό το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Είναι το πρόβλημα παλιό, είναι το πρόβλημα παγκόσμιο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε χώρες αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες. Είναι μια πραγματικότητα που έχει να κάνει με τις διαλυμένες οικογένειες και έχει να κάνει βέβαια και με τα κατώτερα, τα λαϊκότερα στρώματα. Όμως τελικά είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που συμβαίνει σε πολλές οικογένειε οικογένειες ανεξάρτητα οικονομικής κατάστασης ή παιδείας. Είναι πάρα πολλέ οι γυναίκε οι οποίε έχουν υποστεί τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του μια τέτοια εκδήλωση βία. Επομένω γι' αυτό θα πρέπει να τι βοηθήσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε μια σειρά πρωτοβουλειών που να κατατείνουν στον ίδιο σκοπό. Νομική, δικαστική αρρωγή, μέτρα τα οποία θα συγκροτήσουν κάποια καταφύγια, κάποια, κάποια ε, κάποιους οίκους προστασίας αυτών των, ε, ε, αυτών των προσώπων γιατί πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη ζημιά την οποία παθαίνουν τα θύματα τέτοιας επιθετικότητας. Βεβαίως το παίρνει και το θέμα του πόσο κοστίζουν αυτά τα φαινόμενα, γι' αυτό και χρειάζεται μια γενική κινητοποίηση πολιτική και κοινωνική. Πρόκειται περί εξασφάλισης της ανάπτυξης και της ισότητας. Επομένως θα πρέπει με καινούργια μάτια να δούμε την υπόθεση αυτή για να δούμε και τι θα γίνει με τη χρονιά κατά πολέμηση της βίας των γυναικών και πώς θα ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους κατά αυτού του κακού. Σας ευχαριστώ τώρα και το κύριε Μπλίν και Βίτσου. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να ευχαριστήσουμε την Εύα για αυτή την αξιολογική έκθεση. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία μας ε, δίνει μια πάρα πολύ ακριβή εικόνα αυτής της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρόκειται για φαινόμενο που δεν έχει όρια, δεν γνωρίζει σύνορα ή κοινωνικά, γεωγραφικά, οικονομικά. Επομένω, θα πρέπει η κοινωνικα γεωγραφικα οικονομικα Επόμενο θα Επιτροπή να εκπονήσει μια στατική διαδικασία αυτού του φαινομένου και να το κάνει αυτό το γρηγορότερο δυνατόν. Οπότε και με τη σειρά μου να ενθαρρύνω την Κομισιόν να ανλάβει άμεσα δράση γιατί η βία κατά των γυναικών πάει χέρι-χέρι με την σεξουαλική εκμετάλλευση. Ακροτηριασμός γεννητικών οργάνων, λευκή γάμη, είναι κάτι το οποίο υπονομεύει ανέκλητα την υγεία και την ψυχή της γυναίκας. Επομένως θα πρέπει να έχουμε γενικού λειτουργού, να έχουμε δικαστήρια, να έχουμε διοικητικέ αρχέ που να συντονιστούν τόσο να καταπολεμηθεί αυτή η βία κατά των γυναικών. Να ευχαριστήσω επίση και την κυρία Μάλτον γιατί κατέβαλε προσπάθειε για να βοηθήσει τι μη κυβερνητικέ οργανώσει που βοηθάνε στην υπόθεσή μα. Στη σημερινή συγκυρία τη οικονομική κρίση έχουμε ακόμη περισσότερη βία Άρα δεν θα πρέπει με τίποτα να μειωθεί η χρηματοδότηση για την κατέληξη του φαινομένου. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Και. τελευταία θα λάβει το λόγο η κυρία Φασίκοβα. Για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η βία κατά της των την πάτηση των δικαιωμάτων είναι κάτι που μας απασχολεί και πολλά χρόνια και θα πρέπει να σταματήσουμε αυτά τα εγκλήματα το έβρος βίας κατά των γυναικών ε, καλύπτει όλες τις γυναίκες και τις γυναίκες της οικογένειας τους και εκτός ε, τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν τη βία αυτή είναι θύματα, έστω και έμεσα θύματα και θα πρέπει λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τις γυναίκες αυτές και τα παιδιά που είναι θύματα της ε, οικογενειακής βίας. Ε, επίσης η προστασία των πιο ηλικιωμένων γυναικών είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη. Είναι περιορισμένη πολλές φορές η οικονομική της δυνατότητα, ε, η προσωπική της δυνατότητα. Επίσης το εμπόριο των γυναικών είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν πιο αποτελεσματικές κυρώσεις. Ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι τα εγκλήματα θα πρέπει να φροντίσουμε να αποτραπούν στο μέλλον αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Ευχαριστώ. Και τώρα περνάμε στις παρεμβάσεις Catch the Eye. Υπάρχουν 15 συναδελφοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Είναι σημαντικό το θέμα, γι' αυτό υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση. Κερδίσαμε λίγο χρόνο γιατί λείπαν κάποιοι συνάδελφοι. Θα δώσω το λόγο παρακάτω στην αδερφή. Δεν θέλω να, να αναφέρω τους συναδέλφους που δεν μπορούν να ξαναμιλήσουν γιατί ήδη μίλησαν. Ούτως ή άλλως επιτρέπουμε σε πολύ περισσότερους να πάρουν το λόγο κατ' εξαίρεση. Ο κύριος Κέλλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο πράγματα θέλω να τονίσω. Τη βία, ε, θέλω να μιλήσω για τη βία εναντίον των γυναικών και δεύτερον για την θέση των ανδρών ε, που εργάζονται σε ξενοδοχεία. Η βία είναι απαράδεκτη. Ε, χρειάζεται ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ε, μεταξύ των νεαρών ανδρών να διαχειρίζονται το θυμό τους για να αντιμετωπίζουν σωστά τις γυναίκες. Ε, συχνά οι ιδέες που έχουν για τις γυναίκες είναι, βασίζονται σε κάποια ταμπού. Επίσης θέλω να μιλήσω για το ρόλο των ανδρών. Στα ξενοδοχεία, ως πορτιέρδε κτλ. Ε, υπάρχει ζευγά, ε, μία κοπέλα μάλλον, η οποία σκοτώθηκε ε, στο Μαυρίκιο, στο ξενοδοχείο της, όταν κάποιος μπήκε μέσα στο δωμάτιο της για να την κλέψει. Θα πρέπει να δούμε τους κινδύνους, τις πιθανότητες ε, την πρόσβαση που έχουν οι άνδρες ε, στα δωμάτια γυναικών επίσης. Ε, γιατί από εκεί απορρέουν διάφοροι κίνδυνοι. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που σας έχουμε δώσει. Ήμουν ήδη γενναιόδωρος, τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Ταραμπέλα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφο, χαιρετίζω την έκθεση της κυρίας Βέτσεν ε, που τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε όλες τις μορφές βίας ως ε, εγκλήματα του ποινικού δικαίου. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αποτελείται από διάφορους πολιτισμούς και κουλτούρες, αλλά σε ό,τι αφορά την βία θέλω να μεταχειριστούμε διαφορετικά τα θύματα. Παραδείγματο χάρη, ε, ο βιασμό. Παντού είναι αδίκημα του ποινικού δικαίου, αλλά δεν τον αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο παντού. Ε, Παραδείγματο χάρη, στη Λετωνία δεν νοείται ότι σε βιάζει ο άντρα σου. Στη Μάλτα, ε, ο βιασμό άντρα από άντρα δεν υπάρχει. Και στη Σλοβακία, το να βιάσει κανεί ε, με ένα αντικείμενο, αυτό δεν νοείται. συχνά ζωέ καταστρέφονται, ε, συχνά υποτιμούμε τη σημασία των εγκλημάτων και το, τα βάσανα των θυμάτων. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν να φτιάξει πολύ γρήγορα ένα οδικό χάρτη ε, για να καταπολεμήσουμε όλες τις μορφές της βίας πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είδαμε στη συζήτηση ξεκάθαρα ότι η βία κατά των γυναικών είναι πραγματικά μια ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει ότι και τα παιδιά είναι πολλές φορές έμεσα θύματα της βίας κατά των γυναικών, μπορούν να είναι και άμεσα ε, θύματα, γιατί ο κύριος λόγος για την γέννηση ε, νεκρών εμβριών, οι αποβολές είναι πολλές φορές η βία κατά της μητέρας και δεν πρέπει να μην ξεχνάμε το θέμα της ακροτοκτορισμού των ε, γενικών οργάνων, το εμπόριο των γυναικών κλπ. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή η έκθεση αυτή γιατί είδαμε ότι η ισοτιμία επίσης πλήττεται από τη βία κατά των γυναικών αλλά και γιατί έχουμε τώρα τη δυνατότητα μέσα στη του Λασσαβόνας να προχωρήσουμε σε μια οδηγία, να έχουμε κοινό νομικό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γιατί εδώ έχουμε ένα διευρωπαϊκό ε, φαινόμενο. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Βέρτμαν έχει το λόγο. Ένα λεπτό. Η βία κατά των έχει πολλές ε, μορφές και εξακολουθεί να είναι ένα διεθνές φαινόμενο που δεν ελέγχεται από την παγκόσμια κοινωνία. Η βία κατά των σημαίνει υγεία, ασφάλεια των, και αξιοπρέπεια των θυμάτων να πλήττεται. Εκτός από το ότι η βία κατά των ιερικών είναι και κοινωνικό φαινόμενο, εάν κανείς ε, σκεφτεί παραδείγματος χάρη τα φαινόμενα στο τομέα της υγείας και της δικαιοσύνης. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στα σπίτια τους. Σε περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει το θέμα της οικογενειακής βίας. Η βία κατά των γυναικών δεν είναι παράπτωμα. Η διάκριση κατά των γυναικών θα, η, η, η σύμβαση για διάκριση των γυναικών θα πρέπει να υπογραφεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Νικολάσικ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νικολάση, όχι Μικολάση. Ευχαριστώ. Η βία αυτή έχει μακρόπνοες και καταστρεπτικές συνέπειες για την οικογένεια και για την κοινωνία και θα πρέπει να καταδικαστεί ε, όταν στρέφεται αντίον των γυναικών και των παιδιών. Η οικιακή βία μάλλον είναι ο βασικός λόγος για τις αυθόρμητες αποβολές. Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας στα πλαίσια του ποινικού δικαίου για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα εγκλήματα. Θα ήθελα να μιλήσω για την ε, ύψιστη ανάγκη προστασίας των γυναικών και των φτωχών ε, γυναικών οι οποίες γίνονται ε, εξ ανάγκης παρένθετες μητέρες για λόγους οικονομικούς. Ξεχνάμε εδώ ότι με αυτόν τον τρόπο ε, υπάρχει μια απαγόρευση ε, κατά του της εμπορίας ανθρωπίνων οργάτων. Ε, υπάρχει μια εμπορία μέσω των παρένθετων μητέρων. Εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και σώματος. Η κυρία Μικολάσικ τώρα. Ευχαριστώ. Παρόλο που είναι συχνό φαινόμενο βία κατά των γυναικών, δεν υπάρχουν κυρώες γι' αυτό. Πολλές φορές υπάρχουν για άτομα που βρίσκονται σε ε, κατάσταση διαμάχης σε ορισμένες φορές οι χώρες τους ή και άλλες χώρες. Υπάρχουν χώρες που έχουν προβλήματα με τη βία κατά των γυναικών, την πορνεία, την, ε, τον ακροτισμό των γεννητικών οργάνων κλπ. Και επίσης και τα κορίτσια είναι θύματα βία συχνά και θα πρέπει αυτό τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να έχουν πλήρη στατιστικά στοιχεία, να έχουν πλήρη παρουσίαση των ε, συμβενών αυτών όσον αφορά την ε, σεξουαλική βία για να μπορέσουν έτσι να υιοθετήσουν τα κατάλληλα μέτρα κατά των φαινομένων αυτών. Θα πρέπει και στο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των ε, φίλων να δράσουμε επίσης. Ε, ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Νίκολαη, βουλευτής Νίκολαη. Mulțumesc și eu, domnule președinte. În calitatea mea de raportor din umbră doresc să... Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Ως ε, σκιώδη συγγήτρια θα ήθελα να ευχαριστήσω την συγγήτρια και να τη συγχαρώ για το έργο της. Θα πρέπει νομίζω να απομακρυνθούμε από την τυπική εξέταση του θέματος γιατί χωρίς ε, συνεπή ε, αντιμετώπιση και χωρίς ε, οργανωμένη αντιμετώπιση αυτών των ε, εγκλημάτων δεν μπορούμε, δεν αξίζει τον κόπο να συζητάμε. Το οικονομικό κόστος της βίας κατά των γυναικών δεν έχει εξεταστεί μέχρι στιγμής σοβαρά. Αλλά ακόμα και πριν από την έκθεση Έλειπαν πάρα πολλά στοιχεία σχετικά. Παρ' όλα αυτά πιστεύουμε ιδίω στην σήμερα ημέρα που έχουμε την οικονομική ε, και χρηματοπιστική κρίση το κόστος της βίας κατά των γυναικών ε, είναι ζημιά εκατομμυρίων. Θα πρέπει λοιπόν όχι μόνο με οικονομικά αλλά και με πολιτικά μέτρα να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Μόρβα, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την εισηγήτρια. Συνεργαστήκαμε και είμαι πάρα πολύ περήφανη, διότι πριν από 18 χρόνια εγώ έγραψα ε, στη χώρα μου το πρώτο μας κείμενο που είχε ως θέμα αυτό το ίδιο πρόβλημα. Όμως, ακόμα πολλά από να γίνουν στη χώρα μας για το πρόβλημα αυτό. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να έχουμε ίδια νομοθετική ρύθμιση σε όλα τα κράτη. Όμως μπορούμε να έχουμε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο και έτσι αποτελεσματικά να βοηθάει στην πρόληψη, στην αρρωγή των πάθουσών ε, και ε, είναι δυνατόν κύριε Πίτροπε να έχουμε κάποιον έλογο τρόπο διάθεση τέτοιων κονδυλίων, βοηθήσουν κυβερνήσεις να προσφεύγουν εύκολα στις ε, αρχές, στα θύματα. Πάντως και σε Βουδαπέστη και στο Άμστερνταμ και παντού είναι πάρα πολλές οι γυναίκες που πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, σπρώχνονται στην πορνεία. Και επομένω θα πρέπει κάτι να κάνουν κυβερνήσει για να τι βοηθήσουν. Ευχαριστώ με εμεί, λέει ο πρόεδρο, και δίνει τον λόγο στον κύριο Λούαν. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν φαίνεται από την έκθεση αυτή ότι πρέπει να καταβάλουμε διπλές προσπάθειες για να αντιμετωπίσουμε και να καταστήλουμε τη βία κατά των γυναικών. Και εδώ και γενικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπήρου σε όλες τις χώρες που υπάρχει αυτού του τύπου η βία θα πρέπει να ε, αντιδράσουμε τα άτομα αυτά έχουν ψυχολογικά προβλήματα και πολλές φορές τα ψυχολογικά προβλήματα οδηγούν στη βία. Θα πρέπει οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεργαστούν. Θα πρέπει να κατονομάσουμε το φαινόμενο αυτό, θα πρέπει να καταγράψουμε το φαινόμενο αυτό. Και μέσα στα πράσια του προγράμματος της ΟΧΡΟΛΜΗΣ θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πτυχές. Βέβαια, αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να τύχουν και οικονομική ενίσχυση και το κατάλληλο πλαίσιο γι' αυτό θα ήταν το πρόγραμμα δράση. Δάφνη. Δάφνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όταν πρόκειται για θέματα ισότητας, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πραγματικά η πρώτη στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Είναι ακριβό αυτό βέβαια. Η έκθεση λέει ότι κοστίζει 33 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο το αποτέλεσμα της βίας. Και γι' αυτό ε, μπορούμε πραγματικά να κάνουμε να σιωπήσουν εκείνους που θεωρούν ότι ο κατάλογος αυτός των μέτρων είναι πολύ ακριβός, Αλλά Χρειάζεται όμως και κάνουμε οικονομίες. Εκπαίδευση των αστυνομικών αρχών, δικαστικών αρχών κλπ. Όλα αυτά τα λέει η έκθεση της κυρίας Βέσνα και θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Ένα προβληματάκι όμως θα ήθελα να τονίσω. Θα πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην βία στον τόπο εργασία. Γιατί εκεί θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στη διατύπωση. Ευχαριστώ. Και τώρα... Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ρόιτοβα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε φορά που στα ΜΜΕ βλέπουμε ένα θύμα οικιακής βίας, γυναίκα ή παιδί, διερωτώμαστε πώς είναι δυνατόν το περιβάλλον τους να το αγνοούσε τόσο καιρό. Θα πρέπει, λοιπόν, η στρατηγική που ανήκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να περιλαμβάνει συγκεκριμένους μηχανισμούς για τον εντοπισμό ε, του προβλήματος ήδη στα ιατρικά ε, ιδρύματα και στις κοινωνικές υπηρεσίες, ούτως ώστε να βοηθήσουμε αμέσως τα θύματα. Χρειάζονται επίσης αυστηρές ε, κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης κάποιων η χρησιμοποίηση με διαστρεβλωμένο τρόπο ε, κάποιων θρησκευτικών τελετουργικών, ας πούμε, ε, ούτως ώστε να σταματήσουμε τη βία αντίον των γυναικών, τον ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων. Θα πρέπει να έχουν επίσης να προβλέψουμε ε, νομική βοήθεια και πλαισίωση των γυναικών. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση και σε καμία περίπτωση δεν θα είμαι κατά του εκτιμώντας J. ή μάλλον δεν θα το ψηφίσω, διορθώνει η ομιλήτρια, γιατί υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα γιατί, ανάμεσα στη σχέση παιδιού και μητέρα. Τώρα, η κυρία Μάλστρομ έχει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, σας ευχαριστώ για την πολύ σημαντική συζήτηση αυτή για ένα θέμα που Πολλούς από εμά ενδιαφέρει φυσικά. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη σημαντική της έκδοση και τους κοιόδης εισηγητές επίσης. Όπως σας είπα και στην εισαγωγή μου, ετοιμάζουμε διάφορα μέτρα για το θέμα αυτό, το πακέτο των δικαιωμάτων των θυμάτων που είναι πολύ σημαντικό και θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα. Έχουμε επίσης την πολιτική ποιότητα για την αφύπνιση, την συντοπίση του κοινού και επίσης θα δούμε και την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την οικιακή βία, ούτω ώστε να την προτείνουμε στο Συμβούλιο όταν είναι έτοιμη και να γίνει προς υπογράφων μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εφαρμοστεί εκεί που έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν άλλες δύο προτάσεις που έχουμε υιοθετήσει ή μάλλον εσείς έχετε υιοθετήσει. Την οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ε, περιλαμβάνει πολλά προληπτικά μέτρα, αλλά και υποστήριξη για τα θύματα, γυναίκες και παιδιά, σε περίπτωση που είναι θύματα σεξουαλικής βίας ή εμπορίας. Επίσης, ε, στο πακέτο για το άσυλο υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για ευπαθείς ανθρώπους ε, στα πλαίσια της διαδικασίας ασύλου, παραδείγματος χάρη γυναίκες, όταν έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής βίας. Το πρόβλημα, όπως είπατε, τεράστιο και είναι ντροπή που γυναίκες και κορίτσια στην Ευρωπαϊκή Ένωση φοβούνται ε, καθημερινά. Φοβούνται τη βία, φοβούνται το βιασμό, φοβούνται σεξουαλική εκμετάλλευση και φοβούνται ανθρώπους που θα έπρεπε κανονικά να τους ε, εμπιστεύονται περισσότερο, τους συζύγους, τους συντρόφους κτλ. Πρέπει να δράσουμε και να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Είναι ε, μία από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, υπάρχουν και λίγοι, αλλά γενναίοι άντρε που συνεισέφεραν. Γιατί το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τι γυναίκε, είναι ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα υπάρξουν αποτελέσματα μόνο αν συνεργαστούμε άντρε και γυναίκε για να καταπολεμήσουμε το φρικτό αυτό φαινόμενο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη όπου οι γυναίκε και τα κορίτσια δεν θα αισθάνονται τη βία στο πετσί του γιατί ανήκουν σε λάθο φίλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε και τώρα να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σβένσον, την εισηγήτρια. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Σβένσον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίση του συναδέλφου για την αποφασιστικότητα που κατέδειξα. Θα πρέπει πραγματικά να καταπολεμήσουμε αυτή τη βία. Θα ήθελα να πω προ την Κομισιόν ότι εμείς περιμένουμε τη δέσμη για τα θύματα για να μπορέσουν να υποστηριχτούν περισσότερο τα θύματα. Χρειαζόμαστε όμως και μια οδηγία για την καταπολέμηση της ίδιας της βίας. Δεν θα πρέπει να συμφωνεί κανένας με κάθε λέξη της έκθεσης. Αρκεί όμως να πει κανένας ναι για να αποσταλεί ένα έντονο μήνυμα προς την Κομισιόν ότι χρειαζόμαστε μια οδηγία. Είναι σημαντικό να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές κάτω αυτές τις προϋποθέσεις ότι δεν πρέπει να ντρέπονται και λέγοντας ναι προς την έκθεση θα καταδείξουμε ότι ε, εκείνοι που σφάλουν είναι οι θύτες, όχι τα θύματα. Δεν πρέπει να ντρέπονται τα θύματα. Θέλω επίσης να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες επέζησαν με τη βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, με την εργασία των ε, οργανώσεων των γυναικών. Είναι σημαντικό να μην έχουν εκείνοι μόνοι τους την ευθύνη για την ε, επέμβαση στην περίπτωση που οι γυναίκες αυτές υποφέρουν. Θα πρέπει να πούμε ξεκάθαρα ότι υπάρχει υποστήριξη για αυτές τις γυναίκες. Και θα πρέπει επίσης να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να καταδείξουμε ότι υπάρχει πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο ε, υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ομάδα που απειλείται. Όλες οι κοινωνικές ε, ομάδες απειλούνται και παρακαλώ τους συναδέλφους ας στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν είναι αποδεκτό γυναίκες να είναι αναγκασμένες να ζουν κάτω από τέτοιους όρους. Οι γυναίκες μπορούν να δημιουργήσουν καλύτερη ζωή για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους εφόσον έχουν τη δική μας υποστηρίξη. Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά τους συναδέλφους για την αποφασιστικότητα. Από κοινού θα το καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και Ξέρετε είμαι θρήσκο, οπότε θα ήθελα κάτι να προσθέσω. Από πλευρά χριστιανικής, από πλευρά χριστιανικού ανθρωπισμού. Τι γυναίκα την έπλασε ο Θεός. Επομένω και γι' αυτό το λόγο δεν έδωνε κάνει να επιτρέψει η βία που να ασκείται κατά αυτή. Οπότε αύριο θα τελεστεί η ψηφοφορία κάποια στιγμή μετά την μεσημβρία. Σας ευχαριστώ.